Δεν βλέπω να στέκανε στο λόγο. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά. Ενημερώσει. Ανακοινώσει. Οι κύριοι Αθανάσιος Παφίλης και Αθανάσιος Πλεύρης μου κοινοποίησαν ότι θέτουν πέρας στην βουλευτική τους εντολή από τις 14 Οκτωβρίου 2009 λόγω της εκλογής τους στην, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Ελλήνων. Καταγράφω τη δήλωση αυτή και σημειώνω την χειρία των σχετικών εδρών από τις 14 Οκτωβρίου 2009, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 2 της πράξης που αφορά την εκλογή των νόμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, άμεση καθολική ψηφοφορία και δυνάμει το άρθρο 4, παράγραφος 4 του κανονισμού. Οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας μου ανακοίνωσαν την εκλογή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των εξή. Του Σπυρίδωνος Δανέλη, που αντικαθιστά τον κύριο Γιώργο Παπκοσταντίνου. Από 8 Οκτωβρίου 2009. Του κυρίου Χαράλαμπου Αγκουράκη που αντικαθιστά τον κύριο Αθανάσιο Παφίλη από 14 Οκτωβρίου 2009. του κυρίου Νικολάου Σαλαβράκου που αντικαθιστά τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη από 14 Οκτωβρίου 2009. Καλωσορίζω τους νέους συναδέλφους οι οποίοι είναι εδώ παρόντες. και υπενθυμίζω ότι η δυνάμη του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού όσο δεν έχει επαληθευθεί η εντολή τους και όσο δεν έχει κριθεί ενδεχόμενη ένσταση και υπό τον όρο ότι έχουν εκ προημίου ε, καταθέσει τις δηλώσεις ότι δεν ε, ασκούν ασυμβίβαστο με το κοινοβουλευτικό αξίωμα έργο ή